Good evening, with your permission. Καλησπέρα σας. Με την άδειά σας θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, δηλαδή τα ουγγρικά. Θα ακούσουμε τώρα δηλώσεις του Συμβουλίου Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την βία στην ε, λαοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Πρώτα, η κυρία Σεσίλια Βάλστρουμ, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ την Σουηδική. Κύριε Επίτροπε, κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, η Προεδρία θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα της σημερινής συζήτησης. Βαριές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βαριές περιπτώσεις βίας και γενετήσιας βίας σε βάρος των αμάχων. Έχουμε τονίσει κατά επανάληψη ότι ένας αριθμός ενόπλων ομάδων δραστηριοποιούνται στην χώρα αυτή και υποστηρίζονται και από ένα δίκτυο το οποίο εν μέρη είναι εγκατεστημένο στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω για πόσα χρόνια εμπλέκεται και δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κονγκό και στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών για πολύ καιρό προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα στην περιοχή αυτή. Είναι σημαντικό η εμπλοκή αυτή να συνεχιστεί και στον πολιτικό τομέα και στον τομέα της αναπτυξιακή συνεργασία για την οποία θα μιλήσω. Η υποστήριξη αυτή εκφράζεται και με τον τρόπο ότι ο πρώτος είπατος εκπρόσωπο για την περιοχή αυτή και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών ήδη ορίστηκε το 1999. Δημιουργήθηκαν μηχανισμοί για παράδειγμα το πρόγραμμα Artemis στην περιοχή Ιτούρη, συνεργασία με το 2006 με τις ε, δυνάμεις της Αφρικανικής Ενότητας, υπήρξε μεταρρύθμιση των ε, στρατιωτικών δυνάμεων και των αστυνομικών δυνάμεων. Τώρα υπάρχουν ορισμένες καλές ειδήσει. Οι διπλωματικές διασυνδέσεις με το Κονγκό και τη Ρουάντα, οι ε, διπλωματικές σχέσεις δηλαδή, έχουν επαναληφθεί. Και αυτό είναι ικανοποιητικό. Το 2008 και 2009 οι περισσότερες ένοπλες δυνάμεις υπέγραψαν συμφωνίε ειρήνη που πρέπει τώρα να τηρηθούν. Βέβαια η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ασταθής. Πολλές ένοπλες ομάδε στα ανατολικά τη χώρα αυτή δεν εντάσσονται στι τακτικέ στρατιωτικές δυνάμεις. Οι στρατιωτικές επιχειρήσει συνεχίζονται κατά των ενόπλων ομάδων, κυρίω τη FTLR και αυτό έχει ω αποτέλεσμα βαριέ απόλυτε μεταξύ των αμάχων καθώς και το γεγονός ότι αναπτύσσονται επιθέσεις κατά του αμύχου πληθυσμού, αμάχου πληθυσμού. Επομένως έχουμε μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου, έχουμε βία, φόνους, σεξουαλικές κακομεταχειρήσεις και δεν μπορεί να υπάρχει μια συνέχιση αυτής της πολιτικής ανοχής που θέσπισε ο πρόεδρος Καμπίλα τον προηγούμενο Ιούλιο και έχουμε φυσικά την παράνομη εκμετάλλευση και καταλήστευση φυσικών πόρων. Είναι πόροι οι οποίοι ανήκουν στο κράτος αλλά και στο λαό και όχι στις ένοπλες ομάδες. Θα πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν την παράνομη αυτή καταλήστευση πόρων που είναι μοναχά προς το συμφέρον των ενόπλων αυτών παρανόμων οργανώσεων. Έχουμε προβλήματα σε επίπεδο εκλογών, εξάλλου έχουμε προβλήματα παραβιάσεων, ατασταλιών, νοθειών, βίας και νοθείας. Πολλαπλά λοιπόν είναι τα προβλήματα στην περιοχή και σαν αποτέλεσμα το Συμβούλιο χρειάστηκε να πάρει μια σκληρή στάση σε ό,τι αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών στο βόρειο και στο νότιο Κίβου. χωρίς καμία εξαίρεση τόνει στο Συμβούλιο ότι θα πρέπει το κράτος να εξασφαλίσει την νομιμότητα και τη σύλληψη όλων αυτών οι οποίοι παρανομούν εις το κυβού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη στην ειρήνη και την ασφάλεια για όλους τους πολίτες της ε, περιοχής και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια που είναι ζωτική σημασία για να εξασφαλίσουμε την ευμάρεια αυτής της χώρας. Όλοι πρέπει να πράξουν τα απαραίτητα ώστε να εξομαλυνθεί η κατάσταση στο Κονγκό και ιδιαίτερα στο Κίβου. Χρειάζεται επίσης να υπάρξουν βελτιώσεις μέσα από οικονομικές και εταιρικές σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην χώρα αυτή. Έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρώπη είναι απόλυτα στεναρή σε σχέση με τις δεσμεύσεις έναντι του δημοκρατικού Δημοκρατικής ε, Δημοκρατίας του Κόγκο. Θα είμαστε σαφείς και θα μιλήσουμε με παρησία για όλες τις παραβιάσεις που λαμβάνει η χώρα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο Κόγκο θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τον ιδιαίτερο ρόλο που έχει διαδραματίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπω στα ερωτήματα και στα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μάλστρομ και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κάρελ Ντεχούχτ για την Κομισιόν. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και μέλη του Κοινοβουλίου, εδώ και ένα, μέλο, ένα χρόνο η κατάσταση της ΓΟΜΑ που πολιορκούτο από τις δυνάμεις του ΚΕΝΤΕΠΕ ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη και δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα για τις αρχές του Κονγκό και τη διεθνή κοινότητα. Τα πάντα έγιναν ανθρωπίνως δυνατά για να αποφύγουμε το χειρότερο και να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα και μεταξύ του, της Δημοκρατίας του Κονγκό και των ενόπλων δυνάμεων. <clears throat> Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο μπορέσαμε να αποτρέψουμε μια έκρηξη βίας που είχε τεράστια αποσταθεροποιητική δυνατότητα στο Κονγκό. Αλλά οι υποκείμενες αιτίες αντιμετωπίστηκαν μονάχα επιφανειακά και με κοντόφθαλμη πολιτική λογική δεν μπορούν να προκύψουν παρά μονάχα λαθασμένες και ελλειπείς λύσης. Η διεθνής κοινότητα το έχει τονίσει αυτό και γι' αυτό ποντάρει σε μια πιο μακροχρόνια και μακρόπνα αντιμετώπιση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να στείλει μια δύναμη για την ενίσχυση των στρατιωτικών αγημάτων που βρίσκονται ήδη στο Κονγκό. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η κατάσταση που είναι πραγματικά αποτρόπαια, όπως είπε και η Human Rights Watch, δεν θα συνεχίσει να αντιμετωπίζεται με σιωπή και χωρίς να αντιλαμβάνεται κανείς την πηγή αυτών των προβλημάτων και χωρίς να υπάρχει προσπάθεια να αντιμετωπιστούν με μόνιμο τρόπο τα προβλήματα αυτά. Αυτό όμως θα απαιτήσει τη συνεργασία όλων των κυβερνήσεων του Κονγκό και της Ρουάντα, της δύναμης του ΟΗΕ και της υπόλοιπης διεθνούς κοινότητας και στη συνέχεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεις αμφιβάλλει ότι η πολιτική και διπλωματική προσέγγιση μεταξύ της Ρουάντα και της Δημοκρατίας του Κονγκό θα είναι θετική για την ασφάλεια και την ισορροπία της περιοχής και θα επιτρέψει, αν υπάρχει καλή θέληση και αυσιομεριές, να καταλήξουμε σε μια ειρηνική συνύπαρξη και σε μια συνεργασία αμοιβαία θετική και για τις δύο χώρες. Αλλά, μόνο τούτο, Όλα αυτά είναι η αρχή ενός μακρού δρόμου εσπαρμένου με δυσκολίες. Το θέμα του FTLR είναι στην καρδιά όλου αυτού του προβλήματος που σίγουρα <clears throat> περιπλέκουν την κατάσταση. Η παράνομη εκμετάλλευση φυσικών πόρων, η έλλειψη προστασίας των μειονοτήτων, η ατιμορροσία σε μια τεράστια ζώνη χωρίς κρατικές οντότητες όπου οι δημόσιες αρχές δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τον έλεγχο της περιοχής και όπου ακόμα και οι εκπρόσωποι των δημοσίων αρχών είναι τμήμα των ένοπλων αντιπαρατηθεμενών ομάδων, δίσκουν τη δυσκολία αυτή. Με τη ε, συμφωνία αυτή κατάφεραν να τροχοποιηθεί οι, οι απαιτήσει του Μκούντα και του mm. ΣΕΝΤΕΝΤΕΠΕ. Και υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μια καλύτερη μορφή ελέγχου στην περιοχή αυτή. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνει με μια ατιμορρησία η οποία παραβιάζει οποιαδήποτε έννοια διεθνούς δικαίου, κάτι το οποίο ούτε η Ρουάντα ούτε το Κονγκό μπορούν να δώσουν σε οποιαδήποτε φατρία. Σήμερα η παρουσία του ΣΕΝΔΕΠΕ σε ένα αναποτελεσματικό στρατό όπου η σπατάλη είναι στην για διάταξη οδηγεί σε έλλειψη αποτελεσματικής δράσης υπάρχουν παράλληλες αλυσίδες εξουσίας και δίκησης στο Κονγκό και υπάρχει έλλειψη πραγματικής πειθαρχία μέσα στην στρατιωτική δίκηση που δεν κάνουν επωφελείς τις δράσεις. Δεν υπάρχει λοιπόν κατάλληλη πλαισίωση των στρατιωτικών δυνάμεων του Κονγκό και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των ρουανδόφωνων μειονοτήτων. Όλα αυτά θα οξύνουν ακόμα περισσότερα τα προβλήματα τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει ήδη και ιδίως τον προηγούμενο χρόνο. Ούτε η Ρουάντα ούτε το Κονγκό είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν υποφελώς τα προβλήματα αυτά. Μέσα σε αυτό το γενικό πλαίσιο τα πράγματα παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. Η ανθρωπιστική κρίση παρατείνεται χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι θα προκύψει κάποια βελτίωση ή ότι θα σταματήσουν ή θα μειωθούν οι αποτρόπες και ομές ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι καταληστεύσεις, οι λαιλασίες, οι βιασμοί, οι φόνοι κτλ. Η έκθεση των ΗΕ και της Human Rights Watch που ανέφερα προηγουμένως μας δείχνουν την τεράστια έκταση αυτών των τραγικών φαινομένων. Είναι γεγονός ότι οι δράσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο να εξουδετερώσουν τη δύναμη των ανταρτών θα πρέπει να προχωρήσουν, αλλά όχι με οποιοδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι οι οποίοι προκύπτουν από τη στρατιωτική δράση για τους άμαχους, τους αθώους αμάχους. Όλα αυτά χρειάζονται καλύτερο σχεδιασμό, μια επανειεράρχηση των προτεραιοτήτων και μεγαλύτερη ικανότητα προστασία των πληθυσμών. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρώτο καθήκον οποιασδήποτε δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δύναμη των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να λειτουργήσει σε ένα πλαίσιο εντολή χωρί αμφισημίε. Είναι πολύ νωρί να ζητήσουμε η δύναμη των Ηνωμένων Εθνών να αποχωρήσει. Αντίθετα, είναι απαραίτητο να παραμείνει επιτοπίω για να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερο κενό εξουσία στο Κόγκο. Τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία είναι απλώ συστηματικά, συμπτωματικά, δείχνουν πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα. Πρέπει επίση να σταματήσει η πολιτική και η οικονομική συνενοχή από την οποία ευνοείται το FDLR στην περιοχή του Κονγκό και σε άλλα μέρη και μεταξύ ακόμα και των κραλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αγώνας του FDLR δεν είναι πολιτικού χαρακτήρα, αλλά εγκληματικός. Και το πρώτο θύμα είναι ο άμαχος πληθυσμός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ω εκ τούτου χρειάζεται μεγαλύτερη στεναρότης έναντι κάθε μορφής λαθρεμπορίου και συγχρόνως θα πρέπει να προχωρήσει ο αφοπλισμός ε, και η επανισωμάτωση των πολιτοφυλακών και χρειάζεται να υπάρξει και μεγαλύτερη ε, διάβια σε ό,τι αφορά την στάση της κογκαλιζικής κυβέρνησης αντί αυτών που δεν είναι κατά ανάγκη εγκληματίες. Όλα αυτά τα προβλήματα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε μια λύση όχι μόνο εκεί στις τοπικές ρίζες της ε, σύγκρουσης αλλά και στις όμορες χώρες. Η συμφωνία της 27ης Μαρτίου θα πρέπει να εφαρμοστεί αλλιώς θα υπάρξει τεράστια ματέωση στο πνεύμα των πληθυσμών της περιοχής. Και αυτό είναι μια παράγραπτη προϋπόθεση ώστε οι προσπάθειες επανάκαμψης οικονομικής και σταθεροποίησης να μπορέσουν να ευδοκιμήσουν. Ο ρόλος της διεθνούς κοινότητας θα είναι πραγματικά χρήσιμος. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στα προβλήματα αυτά της περιοχής του Κιβού, αλλά για όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχει περάσει το Κόγκο. Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση τη καρδιά του προβλήματο και στην ανοικοδόμηση του Κονγκό. Για να γίνει κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο πρώτο να υπάρξει εδραίωση τη δημοκρατία και εδώ αναφέρομαι στι τοπικέ εκλογέ, τι βουλευτικέ και τι προεδρικέ που θα γίνουν το 2011. Είναι στοιχείο τη δημοκρατία οι εκλογέ, αλλά συγχρόνω θα πρέπει να υποστηρίξουμε του θεσμού και τι πολιτικέ δυνάμει. χωρίς μια διαλεκτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης δεν έχουμε ανοιχτό πολιτικό σύστημα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η ανάγκη να εμβαθύνουμε στην καλή διακυβέρνηση. Είναι τόσο μεγάλη η εμβέλεια των προβλημάτων που η δημοκρατία του Κονγκό δεν μπορεί να τα επιτύχει όλα αυτά μόνο του. Χρειάζεται και υποστήριξη όλη τη διεθνού κοινότητα. Αναφέρθηκε και το θέμα τη ατιμορρησία. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα, διότι εδώ πρόκειται για ένα θέμα πολιτική το οποίο διατρέχει όλα τα θέματα της κρατικής παρουσίας στο Κονγκό. Το πρόβλημα είναι ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν με μονομένο τρόπο. Το κράτος δικαίου σημαίνει και μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλισης, πραγματικές πρόοδου στην οικονομική ευκυβερνησία. Είναι τόσο μεγάλες οι προκλήσεις που χρειάζονται μακρόπνοες πολιτικές, αλλά συγχρόνως αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει άλοθη, ώστε οι άμεσες κατεπίγουσες δράσεις να μην γίνουν πραγματικότητα. Αναφέρομαι κυρίω παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη σεξουαλική βία που τονίστηκε από την έκθεση του Κοινοβουλίου. Η πολιτική θέληση παίζει τον καθοριστικό ρόλο και θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την πολιτική ανοχής μηδέν του Πρόεδρου Καμπίλα. Η Κομισιόν έχει πράξει ήδη πολλά για να το βοηθήσει να εφαρμόσει αυτή την πολιτική βοήθεια προ το δικαστικό σύστημα, βοήθεια προ τα θύματα στη δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά είναι απαραίτητο να υπάρξει μια πλέον στενή συνεργασία για τον αγώνα κατά τη σεξουαλική κακοποίηση επιτοπίου μεταξύ των δυνάμεων του Κονγκό και τη Κομισιόν. Να υπάρξει η εδραίωση του δημοκρατικού συστήματο, ευκυβερνησία, πολιτική θέληση. Αυτέ είναι οι βασικέ αρχέ επί των οποίων θα αρθρώσουμε μια εταιρική σχέση ίσων μαζί με το Κονγκό. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα οι πολιτικές ομάδες έχουν το λόγο. Ο κύριος Κάτσμαρκ ε, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κάθε δημοσιογράφος που γράφει για την Αφρική θέλει να ακολουθήσει τα βήματα του, του Τζόζεφ Κόνραντ. Γι' αυτό ε, οι περισσότεροι εστιάζουν στις αρνητικές πτυχές μιας κατάστασης. Γι' αυτό συχνά εκφράζουν επικρίσεις. Ε, και συχνά ε, βλέπουν πάντα τα σκοτεινά φάσματα. Αλλά η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό δεν χρειάζεται να είναι δε και καλά ε, μια φασματόδης χώρα. Είναι μια χώρα που έχει πάρα πολλούς φυσικούς πόρους και είναι μια χώρα που μπορούν οι αρχές να εξασφαλίσουν το καλό του πληθυσμού. Νομίζω ότι η επιτυχία στην περιοχή του, του Κιβού είναι το κλειδί για μια καλή διακυβέρνηση. για δικαιοσύνη και για ειρήνη. Αν δεν προωθηθούν αυτές οι αρχές, τα προβλήματα δεν θα εξαλειφθούν. Θυμάμαι την αισιοδοξία του 2006. Εγώ ήμουν τότε παρατηρητής στις εκλογές και με μεγάλη χαρά τότε είχα διαπιστώσει κάποια θετικά βήματα, αλλά δυστυχώς η αισιοδοξία αυτή ήταν πρώιμη. Γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι. Γιατί δεν βελτιώθηκε η κατάσταση. Το θέμα νομίζω είναι θέμα οικονομικό, θέμα χρημάτων. Μιλήσατε για την παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Μιλήσατε για την αγορά οπλισμού. Νομίζω ότι ο, ο η παράνομη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε οπωσδήποτε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάικλ Κάσμαν για 1,5 λεπτό. Ε, κάποιες ε, δηλώσεις της Κομισιόν με καθησυχάζουν. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Συμφωνώ μαζί σα. Ε, δεν μπορούμε να φύγουμε γιατί θα δημιουργήσουμε κενό. Και αυτό θα είναι κενό πολιτική βούληση και πολιτική ηγεσία για να επιλύσουμε τα προβλήματα. Έχουμε διεθνεί δεσμεύσει. Ε, να προωθήσουμε το κράτο δικαίου. Θα ήθελα να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα. Ο, η σύγκρουση ξεκίνησε από το 98 και πάνω από 5,5 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Άμεσα ή έμεσα 45.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μήνα. Επίση, υπάρχουν 1.360.000 εσωτερικά εκτοπισμένοι άνθρωποι που φεύγουν από περιοχέ βία. Ε, Α δώσουμε φωνή σε αυτού που δεν έχουν φωνή. Α δώσουμε φωνή σε αυτού που είναι θύματα. Ε, οι θύτε ε, τη ε, λαϊκή δημοκρατία του, του Κονγκό ε, προωθούν τις απαγωγές, ε, τις καταναγκαστικές στρατολογήσεις, το βιασμό, τη σεξουαλική βία ε, πάσης φύσεως εναντίον παιδιών, ανδρών και γυναικών. Ε, τα παιδιά αυτά, οι γυναίκες και οι άνδρες ταπεινώνονται, βιάζονται και ακροτηριάζονται. Έχει περάσει ο καιρός των ψηφισμάτων. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να πετήσουμε ως διεθνής κοινότητα να σταματήσουν αυτές οι φρικαλαιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν. Δύο λεπτά επόμενος ο μιλητής, ο κύριο Μισελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως ξέρετε πάντα είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γίνονται στο Κονγκό. Ενώ ήταν ελπιδοφόρα η κατάσταση μετά από την προσέγγιση Ρουάντας και Κονγκού, χωρίς την οποία προσέγγιση δεν μπορεί να υπάρξει καμία λύση στην περιοχή του Κιβού και πρέπει να την εδραιώσουμε αυτή την προσέγγιση παρά τις συμφωνίες 23 Μαρτίου που αναφέρθηκαν η κατάσταση στα ανατολικά παραμένει ανησυχητική. Διαπιστώσεις. Πρώτον, όσο το FTLR δεν έχει εξουδετερωθεί θα είναι δύσκολο να ειρηνοποιηθεί το ανατολικό τμήμα του Κονγκό. Δυστυχώς αυτή η περιοχή είναι και το πρώτο θύμα της στρατιωτικής πίεσης του δημο... της Δημοκρατίας του Κονγκό που θέλει να αποκόψει τους εξτρεμιστές από την πηγή χρηματοδότησής τους, κάτι το οποίο οδηγεί σε παράπλευρες ζημίες για τον τοπικό πληθυσμό που πιέζονται και από τις δύο πλευρές. Αυτός ο κίνδυνος ήταν προβλέψιμος και όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος θα έπρεπε από την αρχή να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της δύναμης του ΟΗΕ η οποία ακόμα δεν έχει τους κατάλληλους πόρους για να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις αιτήσει και τις πιέσεις επιτόπου και δεν είναι πάντα άψογη η συμπεριφορά της επιτοπίως. Χρειαζόμαστε μια καλύτερη μορφή συντονισμού επιτοπίως και θα είναι εξάλλου πραγματικά παρακινδυνευμένο να έχουμε κριτικές και ε, αντιμετωπίσεις οι οποίες δαιμονοποιούν την UNMIC, τη δύναμη του ΟΗΕ. Επίσης, το πλαίσιο του πολέμου αυτό δεν μπορεί να δικαιολογήσει την συμπεριφορά των δυνάμεων του Κονγκό. Νομίζω ότι η απόφαση του ΟΗΕ να μην υποστηρίξει πλέον τις δυνάμεις του Κονγκό όταν δεν τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητη. Πρέπει η πολιτική μηδενικής ανοχής του Προέδρου Καμπίλα να χαιρετιστεί, αλλά θα πρέπει να γίνει σεβαστή και να τεθεί στην πράξη. Είναι τέτοια κατάσταση του δικαστικού συστήματος ώστε υπάρχει γενικευμένη εντύπωση ατιμορρησίας στο Κονγκό. Γι' αυτό είναι απαραίτητο η Κομισιόν μας να κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσει την επανικοδόμηση ενός δικαστικού συστήματος και όπως ετώνησε και ο κύριος Επίτροπος αυτό το οποίο χρειάζεται το Κονγκό είναι ένα κράτος δικαίου με πραγματικές εξουσίες γιατί αυτή τη στιγμή λείπουν αυτές οι εξουσίες και δημιουργούν ένα πάρα πολύ αχανές κενό Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Μισελ, η Ιζαμπέλ Ντιουράν έχει το λόγο τώρα. Κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, η κατάσταση στο Κιβού, το είπατε και οι δύο, είναι πολύ ανησυχητική. Παρά την παρουσία 20.000 περίπου, περίπου στρατιωτών της Διεθνούς Δύναμης, οι γυναίκες και οι άμαχοι γενικότερα είναι τα κυριότερα θύματα ακόμη και του στρατού του Κονγκό που βιάζει, τις βιάζει συστηματικά. Πρέπει να το υπεθυμίσουμε αυτό για να τονίσουμε το σκανδαλώδη χαρακτήρα της κατάστασης. Αναρωτιόμαστε αν η λύση δεν είναι χειρότερη από το πρόβλημα. Είναι επίσης προβληματικό να επικρίνουμε χωρίς λόγο τη διεθνή δύναμη η οποία κάνει προσπάθειες να βοηθήσει τον εξαντλημένο πληθυσμό δεν είναι ανάγκη να αναθεωρήσουμε τη δική της εντολή αυτό που χρειάζεται να αναθεωρήσουμε είναι τους όρους με τους οποίους την ασκεί για να μπορέσει έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να καταπολεμήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αρχές του Κονγκό έχουν επίσης βαριά ευθύνη για την ατιμορρησία αυτή κατά των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας. Πρέπει να παραμένουν στα στρατόπεδά τους οι στρατιωτικοί και όχι να κυκλοφορούν γενικότερα παντού. Γιατί έτσι παρεμποδίζεται ο διάλογος και η ειρήνευση που θα ήταν ο μόνος τρόπος για να λυθεί το πρόβλημα. Πάντω, σας επαναλαμβάνω ότι συμμερίζομαι αυτά που είπατε και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ενεργός και λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να αποτελέσει μια ειρηνευτική δύναμη. όλα αυτά νομίζω ότι η δράση της είναι απαραίτητη. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σας είχα πει ότι είχατε μόνο ένα λεπτό. Εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Σαμπίν Λούζιν ε, έχει ένα λεπτό επίσης. Η κατάσταση στο Κονγκό είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει βελτιωθεί παρά την παρουσία δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατάσταση του πληθυσμού, του άμαχου πληθυσμού των γυναικών και των παιδιών στο Κονγκό εξακολουθεί να είναι ήκτρια ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν χιλιάδες άτομα να σκοτωθούν, να βασανιστούν, να βιαστούν και η κυβέρνηση, η στρατιωτική, οι, οι στρατιωτικές δυνάμεις της κυβερνήσεως που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ συμμετέχει σε αυτές τις ομότητες κατά του πληθυσμού. Το 2003 ως το 2006 έχουν τονίσει ότι οι μη κυβερνητικοί φορεί οι οποίοι είχαν παρουσία στο Κονγκό δεν ήταν αποδεκτοί από τον πληθυσμό. Ο Καμπίλα δεν έχει δεχθεί να κάνει καμία συμφωνία με αυτούς τους φορείς. Όλα αυτά συμβαδίζουν με την αναζωπήρωση του πολέμου στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό. Γιατί εμείς υποστηρίζουμε μία από τις μεγαλύτερες ε, βίαιες δυνάμεις στο Κονγκό, την FTLR. Εγώ λοιπόν έχω καταθέσει μαζί με την ομάδα της Γκου ένα ψήφισμα κατά αυτής της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Μέλτσερ από τους μη εγγεγραμμένους. Κύριε Πρόεδρε, η εκδίωξη χιλιάδες ατόμων, χιλιάδες φόνοι, δεκάδες χιλιάδες βιασμών, όλα αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί παρά την παρουσία των δυνάμεων του ΟΗΕ. Πριν από 10 χρόνια ξεκίνησε η επέμβασή μας στο Κονγκό, αλλά τίποτα ακριβώς δεν έχει επιτευχθεί. Η περιοχή αυτή που είναι γεμάτη φυσικούς πόρους υφίσταται εκεί το σύνολο του πληθυσμού, ομότητες και καταδυναστεύσεις από τις ενόπλες ομάδες. Είναι μια σειρά από εγκλήματα τα οποία πολλά από αυτά διαπράττονται από τους στρατιώτες του Κονγκό. Παρά το γεγονός ότι έχουν τεθεί κάποιοι ενώπιον του δικαστηρίου της Χάγης δεν έχει προχωρήσει καθόλου αυτή η διαδικασία οι δημοκρατικές δυνάμεις και την απελευθέρωση της Ρουάντα έχουν εμπλακεί μέσα στην ε, διαμάχη στο Κονγκό. Είναι πραγματικά ανησυχητικό ότι αυτή τη στιγμή υπήρξαν και κατηγορίες κατά των δυνάμεων του ΟΗΕ οι οποίες δεν έχουν συμπεριφερθεί με τον κατάλληλο τρόπο. και πολλές φορές συνδέεται η υποστήριξη του στρατού με μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει η δύναμη του ΟΗΕ να συμπεριφερθεί όπως αρμόζει στις ευρωπαϊκές αξίες. Είναι απαραίτητο λοιπόν εμείς να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά με σαφήνεια και κατά την άποψή μου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πρώτα απ' όλα να συγκεντρώσει την προσοχή της όχι στη μακρινή Αφρική αλλά στις περιοχές των Βαλκανίων και του, και του Καυκάσου όπου λαμβάνουν χώρα και εκεί συγκρούσεις μέσα στη δική μας την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στη μακρινή Αφρική. Ευχαριστώ. Οι άλλοι ομιλητές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κατάσταση στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό είναι αξιοθρύνητη και η επίπτωση της σύγκρουσης στους πληθυσμούς προφανώς είναι πολύ δεινή, είναι τραγική. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τονίσουμε και, στο κοινή, και στην κοινική πρόταση ψηφίσματος. Η βία στο Κονγκό, όπως ε, και άλλου τέτοιου τύπου ε, συγκρούσεις, ε, γεννιούνται από την απληστία. Αλλά επίσης εξαπλώνονται και λόγω φτώχειας, λόγω πολιτικής, ε, νομίζω ότι όλα αυτά είναι ε, τα κλαδιά του δέντρου της ε, φτώχειας και της έλλειψης. Νομίζω αυτό, αυτή είναι η πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε ό,τι αφορά την πολιτική ανάπτυξη στο Κοινοβούλιο. Επίσης, η παρουσία μας σε μια ξένη χώρα υποτίθεται ότι θα πρέπει να μειώνει τη βία και τα προβλήματα σε μια χώρα και όχι να την επαυξάνει. Ε, η δυτική παρουσία ε, των δυτικών ομάδων νομίζω ότι δεν ε, συντείνει σε κάτι τέτοιο. Η ιστορία επίσης μας δείχνει ότι τέτοιου τύπου συγκρούσεις όπως αυτές στο Κονγκό ε, επιλύονται με πολιτικό τρόπο. Ο διάλογος ε, νομίζω ότι είναι μοναδική, ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συγκρούσει. συγκρούσεις. Ε, με την συνθήκη της Λισαβόνας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι μπορεί να δράσει έτσι πολύ πιο δραστήρια ε, και να προωθήσει το διάλογο και να αποτελέσει ένα μεκίνα της ειρήνης. Ευχαριστώ. Κύριε Μίτσελ, 1,5 λεπτό, κυρία Κρέτσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκατομμύρια αμάχων έχουν χάσει τη ζωή τους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στα ανατολικά της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό. Τελικά αυτά τα νέα τα ακούμε ε, με αδιάφορο αυτή, γιατί ε, η συχνότητά τους είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα θύματα είναι παιδιά, ε, κορίτσια, γυναίκες και γενικότερα άμαχοι, καθώς και δημοσιογράφοι η ανθρωπιστική κρίση είναι όλο και πιο έντονη και η κατάσταση της ασφάλειας δεν επιτρέπει πλέον στις ανθρωπιστικές οργανώσεις να παρέμβουν. Χιλιάδες βιασμών παρατηρήθηκαν στο πρώτο τμήμα αυτού του, του τελευταίου μήνα. Πολύ περισσότεροι από ότι την ίδια περίοδο πέρυσι. Και φυσικά αυτές, αυτή η στάση, ας πούμε, ε, οφείλεται στη φτώχεια, οι εξεγερμένοι και ο στρατό επιδίδονται σε τέτοιε δραστηριότητε και δυστυχώ μεγάλη ευθύνη έχουν και τα στρατεύματα του ΟΗΕ στο Κονγκό που κλείνουν τα μάτια σε σοβαρότατε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διρωτηθεί για τον τρόπο με τον οποίο οι ειρηνευτικέ δυνάμει εξυπηρετούν του στόχου τη αποστολή του. Επίση, θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για να σταματήσουμε το ξέπλυμα του χρήματο και το λαθρεμπόριο των διαμαντιών και, των, ε, και του χρυσού. Ε, ξεχνάμε ότι 37.000 τόνοι ε, διοχετεύονται λαθρέως έξω από τη χώρα κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής, η κυρία Σόφι Ιντβέλτα. Eh, θα ήθελα να επανέλθω στον συνάδελφο Μίλλερ, ο οποίος τόνισε ότι θα πρέπει να δώσουμε περιγαλύτερη έμφαση στους γειτονές μας. Αν εξετάσουμε όμως την κατάσταση, το ερώτημα είναι πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα στο Κονγκό. Εγώ σκέφτομαι όμως τις γυναίκες που ήρθαν στο Κονγκό και μας επισκέφθηκαν, για τις οποίες μίλησε και η κυρία Ντυρό, και θα πρέπει να δούμε και τους ανθρώπους και τα βάσανά τους, δεν πρέπει να τους αφήσουμε στην τύχη τους. Εμείς δεν αρκεί να περάσουμε ένα ψήφισμα και να θεωρήσουμε ότι έχουμε λύσει το πρόβλημα. Πρέπει να μπορούμε να κοιτάξουμε αυτές τις γυναίκες με την πικρία τους και την απόγνωσή τους στα μάτια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα με τέτοιο επιφανειακό τρόπο. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτό το ψήφισμα <clears throat> και νομίζω τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε, να προσθέσουμε και την δράση μας στα λόγια μας. Μιλάμε πολλές φορές για βία, για σεξουαλική βία, Αυτά είναι μια ορολογία, ορολογία που δεν δείχνει την ομή πραγματικότητα. Δεν είναι μονάχα η απλή επίθεση κατά ατόμων. Πρόκειται για επιθέσεις κατά μιας ολόκληρης κοινότητας με στόχο να διαραγεί ο ιστός ο συνδετικός μιας κοινότητας. Όχι μονάχα πρέπει να δράσουμε λοιπόν, όχι μονάχα να σταματήσουμε την ατιμορρησία η οποία επικρατεί, όχι μονάχα να καταπραίνουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά να έχουμε και μέσα για να υποστηρίξουμε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσουμε ότι θα δείξουμε αλληλεγγύη με τους λαούς της περιοχής αυτής και να μην τους εγκαταλείψουμε στην τύχη τους. Αυτή είναι η ηθική μας ευθύνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δεν έχω, sorry. Αυτή τη στιγμή που τίθεται το ερώτημα της παράτασης εντολής της δύναμης των Ηνωμένων θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά για το σεβασμό των διεθνών συμβάσεων στην, ε, στο έδαφος του, της δημοκρατικής δημοκρατίας του Κόγκο. Γιατί η κατάσταση επιδεινώνεται συνέχεια. Συνέχεια. Και συνέχεια. Αν εξετάσουμε την κατάσταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η στρατιωτική επιτυχία δεν, έχει κανένα νόημα αν το ανθρωπιστικό κόστος είναι πολύ ψηλό. Και το ανθρωπιστικό κόστος σημαίνει δεινά και πάθη των αμάχων. Νομίζω ότι οι πρόσφατες ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στον πληθυσμό και συνοδεύτηκαν από κολοσιαίες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έκαναν την ανθρωπιστική κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή. Η ατιμορρησία είναι η προϋπόθεση της επανάληψης αυτών των εγκλημάτων. Γι' αυτό ακριβώς, κατά την άποψή μου, η προστασία των αμάχων είναι η πρώτη θα πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διατρανώσει ότι η βία και ιδίω η σεξουαλική βία, καθώς και όλες οι παραβιάσεις που είδαμε στο Κιβού θα πρέπει να σταματήσουν πάρα αυτά καθώς και η κατάσταση ατιμορρησίας. Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής παρακαλώ. Ο κύριος ε, Μπαρνιόεβο Γκαρθία. Ένα λεπτό. Ο κύριος Γιάννης. Ζούμε σε μια τραγική κατάσταση στη δημοκρατική δημοκρατία του Κονγκό. Είναι ένα πεδίο θανάτου, βασανισμού και κακοποίησης του λαού εκεί. Η Μόνουκ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν τον έλεγχο καν της παράνομης ροής πρώτων υλών, διαμαντιών, χρυσού, πετρελαίου κτλ. προς τον έξω κόσμο. Γιατί περνάνε αυτά τα προϊόντα από σκιώδεις επιχειρήσεις που τα νομιμοποιούν στις χώρες μας αυτές και στι Πολιτείε είναι απαραίτητο να ανακόψουμε αυτήν την ροή και αυτό είναι καθήκον τη κυρία Άστον. Με τι ευθύνε που έχει τώρα και την αρμοδιότητα από τη Συνδίκη τη Λισαβόνα και με την υποστήριξη των 27 μπορεί να συντονίσει μία σειρά μέτρων για να αποφύγει να μπορούν οι πολέμαρχοι να ενθυλακώνουν τα κέρδη από αυτέ τι ενέργειε οι οποίε βασίζονται σε παραδιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ, λέγει ο πρόεδρο. Ο επόμενο ομιλητή, 1,5 λεπτό. Η κυρία Ντελβού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι μίλησαν για κατεπίγουσα κατάσταση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα για το Κονγκό. Με βάση τις ε, πρόσφατες ε, εκθέσεις που έχουμε για τα βόρεια ε, και για το νότο του Κιβού λόγω των επιθέσεων στους αμάχους και στις γυναίκες στα παιδιά και στους ηλικιωμένους, νομίζω ότι ε, μας αναγκάζει να κινηθούμε πάρα αυτά. Όλα πρέπει να γίνουν για να εξασφαλιστεί η προστασία των αμάχων πληθυσμών. Η εντολή της Μονίουκ θα πρέπει να παραταθεί βεβαίως, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να αναθεωρηθεί και να ενδυναμωθεί για να σταματήσει η βία. Εδώ και πολλά χρόνια η διεθνής κοινότητα, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οι, κο, οι κογκολέζες γυναίκες ίδιες προσπαθούν εδώ και χρόνια να σταματήσει η χρήση όπλων ε, με σεξουαλικό τρόπο, σεξουαλική βία που συνοδεύεται βέβαια από ατιμορρησία. Χαίρομαι για το γεγονός ότι οι κογκολέζικε αρχές αποφάσισαν να θέσουν τέρμα σε αυτή την ατιμορρησία. Αυτή η πολιτική ε, Τη μηδενικής ανοχή, θα πρέπει να είναι φιλόδοξη και όλοι οι δράστε θα πρέπει να λογοδοτήσουν. Η πολιτική θα πρέπει να είναι ε, αποτελεσματική. Θα πρέπει να αρχίσει ε, στο ποινικό δικαστήριο η πρώτη δίκη των ε, υπευθύνων και θα πρέπει να καταλήξει στον, στη στυλίτευση όλων των υπευθύνων πολύ σύντομα. Όλα αυτά βέβαια προϋποθέσουν, προϋποθέτουν την ενδυνάμωση των κρατικών φορέων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, παιδιών και γυναικών ε, συχνά η αξιοπρέπεια των παιδιών και η αθότητά τους θυσιάζονται ε, λόγω της αδιαφορίας όλων μας. Ευχαριστώ κυρία μου. Και τώρα προχωράμε στη διαδικασία του Catch the Eye. Έχω οκτώ άτομα που θέλουν να μιλήσουν. Έχουμε οκτώ λεπτά. Ένα λεπτό έκαστος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να μιλήσουν και οι 8 αν όλοι τηρήσουν το χρόνο τους. Κύριε Πρόεδρε, η ανθρωπιστική κατάσταση στο Κονγκό και ιδιαίτερα στην ανατολική του περιοχή είναι καταστροφική. Η κατάσταση του πληθυσμού έχει χειροτερεύσει μετά από τη στρατιωτική παρέμβαση που έκαναν από κοινού οι στρατοί του Κονγκό, της Ουγκάντας και της Ρουάντας. Παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και σημειώνονται βιασμοί. Και γενικά όλα αυτά έχουν γίνει πια πράγματα μπανάλ και καθημερινά. Επιθέσεις σημειώνονται ακόμη και κατά των εργαζομένων στις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Οι εκτοπισμένοι είναι, ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδων και 165.000 μόνο συγκεντρώνονται στην ανατολική περιοχή. Ήδη έχουν ταυτιστεί άλλες 150.000 ιδιαίτερα ευαλώτων ατόμων και πρέπει αυτοί να προστατευτούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταραμπέλας. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, όλοι ολώνησαν την τρομερή κατάσταση που ισχύει στο Κονγκό και ιδιαίτερα στο ανατολικό του τμήμα, βιασμοί κλπ. Αλλά αντί να μιλάμε μόνο για αυτό το θέμα, μπορούμε να επισκεφθούμε την ιστοσελίδα της UNICEF για να τα δούμε εκεί αυτά που συμβαίνουν. Σημειώνονται επιθέσεις κατά γυναικών, δολοφονούνται γυναίκες και Αποφεύγονται έτσι οι γεννήσεις νέων πολιτών στο Κονγκό που να αναπτύξουν τη χώρα στο μέλλον. Για να υπάρξει σταθερή ειρήνη πρέπει οπωσδήποτε ο ΙΕ και η κυβέρνηση του Κονγκό να καταπολεμήσουν τις σεξουαλικές αυτές επιθέσεις για να κυριαρχήσει επιτέλους το δίκαιο εκεί. Ευχαριστούμε κύριε Ταράμπελα, η κυρία Ρίστορα. κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Θέλω να τονίσω τη σημασία τη σεξουαλική βία στο ανατολικό τμήμα του Κονγκό. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει ενοφανέ, είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, έχει παλέ διαστάσει, είναι ψυχικά και σωματικά βάσανα των θυμάτων που οδηγούν και στην κοινωνική τους ε, στον κοινωνικό του αποκλεισμό από την κοινότητά του, που είναι ακόμα πιο τραγικό. Οι πολιτικέ του πρόεδρου Καμπίλα αποδίδουν κάποιου καρπού, αλλά μόνο μια συνολική πολιτική θα μπορέσει εν καιρό να αντιμετωπίσει αυτή τη μάστιγα. Ξέρω ότι η Κομισιόν παρεμβαίνει με μια σειρά από και υποστήριξη στον προπολογισμό του Κονγκό, αλλά μπροστά στι τρομερέ μαρτυρίε τι οποίε βλέπουμε, Ίσως θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι γυναίκες, κύριε Επίτροπε, είναι οι κύριοι φορείς ειρήνης και αποκατάστασης σε μια χώρα όπως το Κονγκό, ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους εσείς θα πράξετε περισσότερα και πιο γρήγορα στο Κονγκό. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρος. Ακολουθεί ο κύριος Ρωμέβα Ιρουίδα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σαφής η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταγραφή παραβιάσεων και κακοποίησεων. Θα πρέπει και πάλι να εκφράσουμε τη λύπη μας για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και νέων κοριτσιών στις ανατολικές επαρχίες του Κονγκό. Εγώ θα ήθελα εξ ονομάτων του εαυτού μου και όλων των συναδέλφων να ζητήσω από όλε τι αρμόδιε ε, αρχέ να φέρουν ενώπιον των δικαστηρίων του ε, αυτού που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα και να ζητήσουμε από τα Ηνωμένα Έθνη να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσουν τις επιθέσεις αυτές κατά το αμάχου πληθυσμού στο Ανατολικό Τμήμα της Δημοκρατίας του Κόγκο. Ζητώ από την ε, συνέλευσή μας να ενισχύσει τον αγώνα κατά της ατιμορρησίας και να κάνει σεβαστό το κράτος δικαίου και αναφέρομαι κυρίως στους βιασμούς των γυναικών και των κοριτσιών και το γεγονός ότι υπάρχουν παιδιά στρατιώτες ακόμα στο Κόγκο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Όμπερ Μάιερ το Δεκέμβριο του 2000, τον 2009 υπήρξε μια ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Κονγκό και Ρουάντα που ήταν ελπιδοφόρ. Αυτό ελπίσαμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό το διχασμένο κράτος και τον πληθυσμό του ο βρίσκεται μεταξύ δύο πυρών. Αλλά όλες αυτές οι ενδείξεις της ε, βελτίωσης της κατάστασης στο Κονγκό δεν έχουν τύχει συνέχισης. Τι θα κάνει τώρα η Κομισιόν για να μπορέσει να ενισχύσει την προσέγγιση μεταξύ του Κονγκό και της ε, Ρουάντα σε σχέση με την εντολή του ΟΗΕ. Πολλοί αναφέρθηκαν στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής εντολή στον ΟΗΕ να προστατεύσει τους βασανισμένους, τους κακοποιημένους στο Κονγκό και ιδίως τα παιδιά μια τέτοια εντολή είναι απαραίτητη στον ΟΗΕ και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να περιμένουμε να κάνει κάτι ο ΟΗΕ με μια τόσο περιστοϊκή εντολή. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα όπλα για να προστατεύσει τους κακατατρεγμένου. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής, ο κ. Σίμκο. Είναι ατυχές που τη χριστουγεννιάτικη περίοδο Ξοδεύουμε τις τελευταίες ε, δύο μέρες να συζητάμε βίες περιοχές, Τσετσενία, Αφγανιστάν και Κονγκό. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παράλληλα, ε, η γιορταστική αυτή περίοδος ε, θα πρέπει να μεταδώσει ένα, δίνει, ένα μήνυμα ειρήνης. Όπως είπε σωστά και ο κύριο Μίτσελ, θα πρέπει να γίνουμε οι μεκίνες της ειρήνης. Είναι μια κατάλληλη ευκαιρία για την είπα την εκπρόσωπο, την κυρία Άστον, να βοηθήσει ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση από πίσω τη για να υπάρξει ειρήνη και τάξη ούτω ώστε αυτά τα μέρη να μπορέσουν να ζήσουν πιο ειρηνικά. Μακροπρόθεσμα όμω, η λύση δεν θα έρθει μόνο από την οικονομική βελτίωση αλλά από την εκπαίδευση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στην παιδεία, σωστή παιδεία σε αυτέ τι χώρε, γιατί αυτό είναι ο δρόμο για να πορευτούμε προ την ειρήνη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κύριε Κέλλη, ο κύριος Higgins. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 1960 ο Γενικός Γραμματέας που ήταν Σουηδό ε, του ΟΗΕ τώρα ζήτησε από τα Ιρλανδέζικα στρατεύματα ε, να πάνε στο βελγικό τότε Κονκό ε, και έκανα μια θαυμάσια δουλειά. εγώ ανησυχώ για τη δουλειά που κάνουν τα στρατεύματα του ΟΗΕ. Ε, Μαροκινοί, Πακιστανοί και Ινδοί. Μιλάμε για βία, για βιασμούς. Ε, δεν νομίζω ότι είναι ένδοξες οι πράξεις των στρατευμάτων της Μονίκ. Συμφωνώ με τον κύριο Μίτσελ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει στεναρότητα. Ε, στο τσάτ τα καταφέραμε. Χρειαζόμαστε τους δικούς μας ε, ειρηνοποιούς και εδώ και δεν πρέπει να βασιζόμαστε στον ΟΗΕ. αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα της ευρωπαϊκής απειοκιοκρατίας. είναι θύματα ε, σύγκρουσης μεταξύ φυλών. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Higgins, Ο κύριος Σβένσον. Ένα λεπτό κι αυτός. Ευχαριστώ. Είναι σχεδόν αδύνατον να καταλάβουμε τις φρικόδεις στατιστικές που ακούμε ε, για τις περιοχές αυτές και όμως ξέρουμε ότι είναι αληθείς έχουν την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για τις στοχότερες από τις στοχές ε, χώρες, την υποσαχάρια Αφρική, ε, οι δεσμεύσει θα πρέπει να είναι μικρότερες από ό,τι για τις ε, υπόλοιπες χώρες. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική δύναμη. Ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την πρόοδο και τη διαφθορά, αν θέλουμε να βοηθήσουμε να βελτιωθεί η κατάσταση σε μια χώρα όπου ο πληθυσμό σήμερα ε, έχει βασανιστεί τόσο, τόσο πολύ. Μιλήσαμε για το Αφγανιστάν, Μιλήσαμε για την τρομοκρατία στο Αφγανιστάν, μιλήσαμε για τους Ταλιμπάν. Εδώ έχουμε τώρα έναν άλλο λαό, ο οποίος έχει επίσης ε, βασανιστεί και έχει βασανιστεί πολύ άσχημα. Θα ήθελα να τονίσω εδώ σήμερα ότι έχουμε οργανώσεις που μπορούν να κάνουν κάτι αν υπάρξει κρατική υποστήριξη και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα Έχουμε τελειώσει τη διαδικασία του Catch the Eye. Η κυρία Σεσίλια Μάλστρομ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι μπορούμε να εξαγάγουμε από αυτή τη συζήτηση. Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι για να συνεχίσουμε την παρουσία μας στη Δημοκρατική Δημοκρατία του Κόγκο. Όπως τονίστηκε ήδη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απόλυτα προσφυλωμένη στο να εξασφαλίσει τη μακροχρόνια σταθερότητα, ασφάλεια και ανάπτυξη στο Κόγκο. Ο Επίτροπο κ. Ντεχούχτ μα έδωσε μια σαφέστατη έκθεση για τι προσπάθειε που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή. Τα κράτη-μέλη καθώ και η Κομισιόν κάνουν σαν σύνολο τη μεγαλύτερη συνολική συμβολή στην περιοχή αυτή, η οποία μπορεί να κάνει και τη διαφορά. Σε ό,τι αφορά όμω τη σταθερότητα τη Δημοκρατία του Κονγκό και τη σύνολη περιοχή, είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε αυτή την ασφάλεια. Θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκε διαβίωση, να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να έχουμε μια στεναρή και αυστηρή αντιμετώπιση για τη διαφθορά σε μια κοινωνία που πρέπει να διέπεται από κράτος δικαίου. Όταν, μιλά, όταν ακούμε αυτές τις τρομερές αποτρόπες ιστορίες για σεξουαλική βία από όλες τις εκθέσεις, είναι προφανές ότι αυτό είναι απόλυτα απαράδεκτο και οι δράστες δεν μπορούν να παραμείνουν ελευθερία. Θα πρέπει όλοι να έλυνε να έρθουν ενώπιον των δικαστηρίων και εδώ υπάρχει πραγματική ευθύνη τη διεθνούς κοινότητα να εξασφαλιστεί ότι η πολιτική μηδενική ανοχή του Πρόεδρου Καμπίλα δεν είναι μονάχα λόγια αλλά είναι και πράξη. Ό,τι αφορά <clears throat> το Συμβούλιο, η εντολή της ΚΕΠΑ που υπάρχει αυτή τη στιγμή και η συνέχιση της αποστολής μα το 2009 έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν και να αναχαιτήσουν την σεξουαλική βία. Θα στείλουμε δύο πολυκλαδικές ομάδες στο Κονγκό, οι οποίες έχουν ιδιαίτερους τομείς ειδίκευσης, αντιμετώπιση του εγκλήματος, αντιμετώπιση σεξουαλικής βίας και θα κινηθούν και στο βόρειο και στο νότιο Κινηβού. Θα έχουν μια εντολή που θα καλύπτει όλη τη χώρα και θα μπορέσουν να δράσουν και ξεκινάει τώρα η στελέχωση αυτών των δυνάμεων. Όλα αυτά είναι μονάχα μια σταγόνα εν το ωκεανό. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να έχουμε ειδικευμένο προσωπικό επιτοπίως για να υποστηρίξει την εφαρμογή των διαδικασιών που είναι απαραίτητε για να αντιμετωπιστεί η σεξουαλική βία, ιδίως όταν αυτή η βία ασκείται από στρατιώτε. Θα περάσουμε σε λίγο στο χρόνο ερωτήσεων προς το Συμβούλιο, αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτή είναι και η τελευταία μου παρουσία ως εκπροσώπου του Συμβουλίου, ενώπιόν σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές που ζήσαμε μαζί και τη θερμή σας υποδοχή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας ευχαριστήσουμε κυρία Μάλστρομ γιατί ήταν πολύ επωφελής ε, η συνεργασία μαζί σας. Ε, ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Τεχούχτ από την Κομισιόν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου που παρενέβησαν σε αυτή τη συζήτηση. Δεν θα επανέλθω στις ε, αρχικές μου παρατηρήσεις και παρέμβαση. Τρία πράγματα θέλω να πω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω προγραμμάτων για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Μιλάμε για πολλά προγράμματα και για πολλά λεφτά. Το θέμα όμως είναι τι αποτελεσματικότητα έχουν εάν δεν υπάρχει εταίρος στην πολιτική σκηνή για να μας βοηθήσει. Δεύτερον, να πω κάτι για την εντολή της Μονίκα. Παρότι η Μονίκα μπορεί να δεχθεί κριτικές και να κατακεραυνοθεί για όσα συνέβησαν πρόσφατα, θα ήταν λάθος παρόλα αυτά να απαιτήσουμε να αποχωρήσουμε από την λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Θα ήταν το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια αποσπάσματα από την εντολή όπως υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στις αρχές του 2008. Λέει ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η Μονίκ θα πρέπει από την υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος να λάβει την εντολή με αυτή τη σειρά προτεραιότητας να συνεργαστεί σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση του Κονγκό, ούτω ώστε πρώτον να προστατεύσει τους ε, πολίτες, ε, το προσωπικό του ΟΗΕ, τις εγκαταστάσεις του, να προστατεύσει τους αμάχους και τους ε, εργαζόμενους ανθρωπιστικές οργανώσεις, να σταματήσει η βία και η βία που προκύπτει από οποιοδήποτε από τους εμπλεκόμενους στην σύγκρουση. Μια άλλη παράγραφος, στην παράγραφο G Μιλάμε για τις συντονισμένες επιχειρήσεις. Εκεί λέμε ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις με το στρατό, με τις ενσωματωμένες ταξιαρχίες που υπάρχουν στα ανατολικά της λαϊκής δημοκρατίας του Κονγκό και που υποστηρίζουν επιχειρήσεις ε, που από κοινού σχεδιάζονται με αυτές τις ταξιαρχίες, ε, με τη διεθνή κοινότητα, με σκοπό την αποκατάσταση του κράτους δικαίου κτλ. Η εντολή είναι σαφής λοιπόν, το βλέπετε. Αυτό που θα πρέπει να ζητήσουμε είναι τους κανόνες εμπλοκής. Και αυτό που θα πρέπει να κάνει η Μονίκ θα πρέπει να εξετάσει τους δικούς της κανόνες εμπλοκής. Γιατί εκείνη θα πρέπει να αποφασίσει πώς θα προχωρήσει. Τέλος, υπάρχουν πολλές επικρίσεις για την διεθνή ποινική δικαιοσύνη. Ορισμένοι λένε αυτό είναι συμβατό τώρα με την πολιτική. Μπορούμε να έχουμε από τη μία το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και από την άλλη μια σωστή πολιτική διαχείριση μιας κρίσης. Σωστό το ερώτημα. Στο Κονγκό όμως δίδεται η απάντηση επιτόπου. Επιτρέψαμε ο Μπόσκο και ο Ταγκάντα να αναλάβουν τη σκητάλη από το CNDP και τον Κούντα. Παρότι υπάρχει ε, ένταλμα σύλληψης του Μπόσκου και του Ταγκάντα. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ή θα διαχειριστούμε πολιτικά την κρίση ή θα υπάρξει διεθνής ποινική δικαιοσύνη. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Εμείς ως Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά η διεθνής ποινική δικαιοσύνη. Θα πρέπει να λειτουργήσει σωστά. σωστα η διεθνή κύριε Ντεχούχτ. Έχουμε λάβει έξι προτάσεις για, από έξι ομιλητές ψηφίσματο, συγγνώμη. Ε, τέλειωσε η συζήτηση και θα ψηφίσουμε αύριο.